του EDF λαμβάνοντας υπόψη την διοργανική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση, ε, μία ακόμη έκθεση του συναδέλφου κυρίου Τυρολιά με θέμα σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Monsieur le Président, chers collègues, l'actuelle Της συμφωνίας η οποία είχε επιτευχθεί ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η συμφωνία αυτή λύγει στο τέλος του έτους. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και να λάβουμε υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών μπορούν να έχουν επιπτώσεις και με βάση τις κλιματικές αλλαγές. Πριν λοιπόν καταδικάσουμε τα υπερπόντια εδάφη, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Υπάρχουν ε, ιδιαιτερότητες και τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα διατρέχουν μεγάλους κινδύνους μέσα στα πλαίσια της αηφορίας. Γι' αυτό χρειάζεται ανανέωση της συμφωνίας για το 14-20 μέσα στα πλαίσια μιας νέας εταιρικής σχέσης αυτή η ε, συμφωνία προετοιμάστηκε πολύ καλά ήδη από το 2008 που εκδόθηκε μια πράσινη βίβλος καθώς και εδώ και δύο χρόνια ολοκληρώθηκε η διαδικασία και γι' αυτό θα ε, και γι' αυτό είχαμε διοργανώσει και μία ακρόαση πέρσι το Σεπτέμβριο. Τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα θα πρέπει να την χάνουν ειδική προσέγγιση για τη μείωση της φτώχειας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Ορισμένα σημεία όμως θα πρέπει να φύγουν ιδιαίτερα για να στραφούμε προς το μέλλον. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες. Ο πρώτος στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υπερποντίων εδαφών και χωρών. Θα πρέπει να έχουν επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αρπούν στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, για να ε, μπορέσουμε να κινηθούμε σε επίπεδο επιχειρήσεων θα πρέπει να ανταποκριθούμε για τη βιωσιμότητά τους. Και θέλουμε να προωθήσουμε αυτές τις δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε η εμπορική πολιτική της Ένωσης οδήγησε σε μία διάβρωση των προτιμησιακών δασμών, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός με τις τρίτες χώρες. Τέλος, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη επαρκώς τους κανόνες προέλευσης για τις επιχειρήσεις ε, και υπάρχει καλύτερη μεταχείριση του Μαυρικίου και των Σεϊχελών. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα υπερπόντια εδάφη. Ένα άλλο σημείο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε το 11 ετά να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και θέματα δημόσιας διαχείρισης για να έχουμε σωστή χρήση του ΕΤΑ στα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα. Τέλος, να σταματήσω λέει ο κύριος Τυρολιά. Εντάξει, σταματώ. Ε, διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Πατράου Νέβες Μαρία Ντοσέου. Ευχαριστώ. Ο ορισμός σωστών και δίκαιων συνθήκων θα πρέπει να ισχύει στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή τη διαδικασία σύνθεσης θα πρέπει να πρόκειται για προστιθέμενη αξία που ε, δρά θετικά. Οι χώρες και τα διαμερίσματα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντοχή και να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα με τους εταίρους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την προέλευση προϊόντων, το σήμα προέλευσης, ιδιαίτερα σε συμφωνίες με τρίτες χώρες και να επαναπροσδιοριστεί μια ευρωπαϊκή διαφοροποιημένη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα αυτών των ε, περιοχών στον τομέα των μεταφορών και της αλίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αρνητική διάκριση από πλευράς Επιτροπής. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Ε, ο συνάδελφος κύριος Πόγκα, Μωρίς Πόγκα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και για τη διαδικασία σύνθεσης Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τις σχέσεις μας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή και υπερποντίων χωρών και εδαφών. Χρειάζεται, ε, χρειάζονται ήδη αγορά αυτές οι υπερποντίες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της νέας απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης της Επιτροπής προβάλλεται ένα νέο μέτρο μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης της φτώχειας και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνεργασίας Γι' αυτό στις διάφορες γενικές διευθύνσεις θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει μία μονάδα για τα υπερπόντια εδάφη. Έτσι θα προχωρήσουμε ακόμα καλύτερα. Και τελευταία ομιλήτρια η συνάδελφος κυρία Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι τα υπερπόντια εδάφη και διαμερίσματα έχουν ιδιαίτερα στρατηγική σημασία. Μέσα στα πλαίσια της απόφασης της υπερπόντιας σύνδεσης θα μπορέσουμε να ε, αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την οικονομική ανάπτυξη στο τομέα του τουρισμού και της γεωργίας. Επίσης χρειάζεται η ιδιαίτερη υποστήριξη της αλίας ιδιαίτερα ως προς την καταπολέμηση της παράνομης αλίας και την ε, ε, προάσπιση των παρακτήων περιοχών. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη ολοκλήρωση των περιφερειακών οικονομιών και συνεργασία με τους εταίρους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτών των εδαφών. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος, κυρία Κόνη Χέντεγκάρτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές και πάλι κύριε Τριολιάν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση αυτή και για την ε, θετική υποδοχή της ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε όλες τις πλευρές και το τελικό κείμενο αποτυπώνει την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των υπερπόντιων εδαφών και χωρών. Η σχετική απόφαση λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ποικιλία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι υπερπόντιες περιοχές και τα εδάφη, αλλά και τις ενδεχόμενες ε, προκλήσεις, τις ενδεχόμενες ευκαιρίες και τα ενδεχόμενα προτερήματα που έχουν. Θα ήθελα να πω ότι σε σύγκριση με την σχετική απόφαση του 2001 σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη ενός κεφαλαίου για το περιβάλλον και για την μείωση σχετικών κινδύνων. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω κάποια στοιχεία για τα μεμονωμένα σημεία της έκθεσης σε ό,τι αφορά τα θέματα ανταγωνιστικότητας. Αποτελούν, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα και τους βασικούς στόχους της συνεργασίας μας και σε ό,τι αφορά, ε, μάλλον σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί και η σχετική απόφαση. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ανταγωνιστικότητα σε συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα ζητήματα της απόφασης. Επίσης, περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιλεξιμότητα των χωρών των υπερπόντιων εδαφών για όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κάποιους όρους. Θέλουμε να συμμετέχουν ενεργά σε οριζόντια προγράμματα. Ωστόσο, η σχετική απόφαση δεν μπορεί να παραβιάσει τη σχετική νομική τάξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για, την τους απλούς ε, για απλούς νόμους και απλούς κανόνες σε ό,τι αφορά την παροχή της βοήθειας <coughs> μετά από διαβούλευση με τις επιπόντιες χώρες και εδάφη θα ε, προταθούν οι σχετικές προτάσεις για την οικονομική αρρωγή βάσει του 10% ου ε, πακέτου και των κατευθυντήριων γραμμών. Σε ό,τι αφορά τώρα το εμπόριο και τους κανόνες προέλευσης, η σχετική απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να βελτιωθούν οι όροι για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Βάσει ενός προτιμησιακού συστήματος ε, πρέπει να σας πω ότι οι κανόνες πηγαίνουν ε, ακόμα παραπέρα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, και άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές, στις ε, χώρες και εδάφη να αποκλίνουν επίσης, απλοποιούνται οι κανόνες για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των αλληλευτικών προϊόντων. Είναι Οι κανόνες από το 2017 και μετά εισαγάγουν το σύστημα της αυτοπιστοποίησης σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις απόψεις που εκφράζονται στο ψήφισμα και γι' αυτό ήδη περιλαμβάνονται στο κείμενο της πρότασης. Φυσικά η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων και των διεθνών ενώσεων. Προς το σκοπό αυτό η απόφαση συμπεριλαμβάνει μια διάταξη για τον ορισμό των όρων και των συνθήκων για να υπάρχει καλύτερη σχέση μεταξύ των οικονομικών μέσων και των εταίρων τη ίδιας περιφερειακής ε, ε, ένωσης. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους, ε, τις χώρες που έχουν και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις Κατά το παρελθόν υπήρξε συνεργασία σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης ε, και υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα. Δεδομένης της ε, σημασίας και της επιτυχίας της συνεργασίας φαίνεται ότι συνεχίζονται οι προτάσεις αυτές στην νομοθετική πρόταση θέματα για την υγεία, για παράδειγμα, τα νοσήματα εξακολουθούν να μας απασχολούν και γι' αυτό λοιπόν γίνονται προτάσεις σε ένα γενικό κεφάλαιο που περιλαμβάνει και την απασχόληση και την ελληνική πολιτική. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου θα εμπλακούν στο ετήσιο φόρουμ